με τον πρόεδρο του Συμβουλίου δύο πράξεις στα πλαίσια της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κοινοβουλίου. Θα δημοσιευθούν